παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος, να εγκαταλείψετε ήσυχο την αίθουσα. Η ησυχία παρακαλώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια καλή ευκαιρία για τον Νότιο ε, Κάφκασο και... Ε, Share with you some thoughts regarding... Ε, είμαι μόνιμος εισηγητής και επομένως ανέλαβα και το θέμα της γεωργίας. Το από το ξεκίνημα της ε, ε, ανατολικής εταιρική ε, σχέσης το 2009 η Γεωργία απέδειξε ότι είναι αξιόπιστος εταίρος και έχει πλέον υφάνει σημαντικό και ε, ε, σχέσεις ε, οικονομικές και πολιτικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει άλλες ανάγκες της γεωργίας όπως ας πούμε προστασία από απειλές της εδαφικής δικαιοδότητας κτλ. Η, αυτή η συμφωνία σύνδεση είναι πολύ σημαντική κυρίως δε αν μιλάμε για deep and comprehensive free trade για την περιοχή. Φυσικά είναι απαραίτητο ε, για να εφαρμοστεί μια τέτοια ε, πιο βαθιά συμφωνία θα πρέπει η Γεωργία να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Τον Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησε η διαδικασία σύνδεσης και υπεγράφει τον Ιούλιο ε, τον Ιούνιο. Μετά από την υπογραφή την 27η Ιουνίου και την κύρωση που ακολούθησε από το ε, Κοινοβούλιο της Γεωργίας ισχύει ε, αυτή η συμφωνία από 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Ε, είναι γεγονός ότι η Γεωργία προχώρησε περισσότερο όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις από τους άλλους εταίρους στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης και κατάφερε να άρει όλες τις ε, όλους τους δασμολογικούς ε, φραγμούς και όλα τα κατάλοιπα ε, της προηγούμενης κατάστασης όσον αφορά τους εμπορικούς δεσμούς και νομίζω ότι ελάχιστε είναι οι χώρες που το κατάφεραν αυτό, η Σιγκαπούρη ας πούμε μου έρχεται στο νου. Στην παρούσα κατάσταση λοιπόν Ε, ε, η Γεωργία ε, προχώρησε ικανοποιητικά με τη βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι μέσω της νέας συμφωνίας DCFTA θα, θα συμπεριληφθούν περισσότερα προϊόντα και οπωσδήποτε θα καλυφθεί και η αμοιβαιότητα. Το δεύτερο το οποίο ε, ήθελα ε, να πω είναι κάτι που ισχύει γενικά με τις ε, περιοχές ελεύθερου εμπορίου με τις, ε, με τις οποίες ε, συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει ε, και σε θέματα τα οποία δεν είναι στρίκτου εμπορικά και επομένως μιλάμε και για την στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα. Όλα αυτά τα κεφάλαια καλύπτονται στο DCFTA με την Γεωργία. Ε, μια ειδική διάσταση πολιτικής ε, αφορά ε, μια ειδική πλευρά της συμφωνίας, δηλαδή σαν ένα μέρος της εταιρικής, ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, η ε, Γεωργία έχει πλέον ένα ειδικό καθεστώς σύνδεση όσον αφορά τους οικονομικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επ' αυτής της όσο προβλέπει διάφορες διατάξεις η συμφωνία όσον αφορά εμπορικές πολιτικές της Γεωργίας που σχετίζονται σχετίζονται με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ε, με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει ε, ε, εξυγχρονισμός της οικονομίας, καλύτερη παρουσία των ευρωπαϊκών επενδύσεων στη χώρα κλπ. Όσον αφορά τώρα τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας, αναμένεται ε, το DCFTA να δώσει μεγάλη όθεση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Γεωργίας ε, και ε, τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τις εξαγωγές από τη Γεωργία και όσον αφορά τις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Γεωργία. Επίσης δίνονται νέες ευκαιρίες εμπορίου και εξαγωγών, ανοίγει η πρόσβαση στην αγορά και ε, επίσης ευελπιστούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ανοίξει ο δρόμος ε, για σταθερότητα ε, και ευημερία που είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους των συμφωνιών σύνδεσης με χώρες της Ανατολικής Συμφωνίας. Επομένως, συμφωνούμε με την άποψη και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να προτείνει στην Ολομέλεια να εγκριθεί ε, η συμφωνία. Επίσης, ε, στο συνοδευτικό ψήφισμα υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία θα ήθελα να καταδείξω ως σημαντικά. Το πρώτο αφορά την εφαρμογή της ε, συμφωνίας που είναι βεβαίως κάτι αυτονόητο και το δεύτερο αφορά την ανάγκη να υπογραμμιστεί ε, η δημοκρατική διάσταση στην εφαρμογή της ε, συμφωνίας κυρίως ε, ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να περιοριστεί στο να απαντήσει θετικά ή αρνητικά σε μια τέτοια διαδικασία και ότι θα πρέπει να έχει τακτική ενημέρωση για τις ε, εξελίξεις κυρίως όσον αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας και αυτή θα πρέπει να είναι μια δέσμευση που θα αναλάβει η Επιτροπή επίσης στο ψήφισμα μου, συγγνωμοδότησή μου, συγγνώμη, ε, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη του γενικότερα την εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Επομένω, σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, για την προσοχή σα. Είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει ή διευκρινήσει όσον αφορά αυτήν την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Νομίζω το τελευταίο σημείο που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό για τη διαχείριση όταν θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει. Παρακαλώ, κύριος Μόζα. Ευχαριστώ. Ως κοιόδης για τον Νότιο Κάφκασο από πλευρά σοσιαλιστών, επιβεβαιώνω ότι η Γεωργία είναι πιστός και σταθερός σύμμαχός μας η αναδιαμόρφωση της εσωτερικής της πολιτικής της εσωτερικής πολιτικής έχει λάβει χώρα ε, με την ενθάρρυνση της Ένωσης που την έχει δεχθεί η ηγετική ομάδα της Γεωργίας αυτή η συμφωνία DCFTA θα ενισχύσει αυτή την τάση θα είναι ένα σύγχρονο μέσο για να εξυγχρονιστεί η οικονομία και οι θεσμοί της χώρας για να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες έχουν γίνει θαραλές ε, παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές για να αυξηθεί η πρόσβαση στις αγορές. Περιορισμένες είναι οι ευαισθησίες των δύο πλευρών και με βάσο και τη συζήτηση που κάναμε μόλις τώρα για την Ουκρανία και θα κάνουμε εντός ολίγου για την Μολδαβία η επικύρωση της συμφωνίας σύνδεσης με, την, με τη Γεωργία θα βοηθήσει πολύ το μέλλον και την περαιτέρω εξέλιξη της χώρας. Έχει και πολιτική διάσταση σημαντική και δεν θα μας κοστίσει πολλά. Ολόθερμα λοιπόν υποστηρίζω τον όλοι για το κείμενο που μας παρουσίασε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Α, η Επιτροπή τότε. Α, με συγχωρείτε, θέλετε να πάρετε τον λόγο. Όχι, καλώς. Ο Ιγνάθιο. Καλωσορίζουμε την γνώμη του κύριου Ρένα και τη στήριξη που δίνει σε αυτήν την πολύ σημαντική συμφωνία και με χαρά θα ενημερώνουμε τακτικά το Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της. Ευχαριστώ. Α, με συγχωρείτε. Α, παρακαλώ, παρακαλώ. Από πλευρά της ΚΟΕ συμφωνούμε με εμπορικές συμφωνίες με πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες αλλά υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσον είναι όριμη η Ουκρανία Γεωργία. η Γεωργία με συγχωρείτε και από πλευρά πολιτικής και από πλευρά οικονομικής για το εάν θα προσαρμοστεί στι προδιαγραφέ που έχουμε σε εμπορικές συμφωνίες. Και έχουμε ανησυχίε και σε σχέση με αυτά που συνέβησαν στην Ουκρανία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να είναι γέφυρες για την ειρήνη και όχι μηχανισμοί απομόνωσης της Ρωσίας. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θα εξετάσουμε την τελική μας θέση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ όλοι. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και έγκριση, για τις ερωτήσεις, για το αν και κατά πόσον είναι έτοιμη η Γεωργία. Κατανοητές οι ερωτήσεις, αλλά κατά τη γνώμη μου πρόσφατα η Γεωργία έχει αναπτυχθεί προς πολύ θετική κατεύθυνση, έχει επανέλθει το εμπόριο με τη Ρωσία. Συναντήθηκα πρόσφατα με εκπροσώπους της Γεωργίας και πιστεύουν ότι η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει ε, την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πολύ καλή μας συνεργασία για το θέμα αυτό. Στη βάση αυτή πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Äh, Ευχαριστώ. Διαπιστώνω ότι έκλεισε συζήτηση για το θέμα αυτό. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 29 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα. Και θα το ξαναδούμε το θέμα στο Στρασβούργο είτε στη συνεδρία μα στις 5-6 Νοεμβρίου. Εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα της ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ότι για το θέμα της έγκρισης δεν μπορούν να γίνουν τροπολογίες παρά μόνο τροπολογίες απόρριψης γιατί μπορούμε να πούμε ναι ή όχι. Όχι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερής διάταξης. Το οποίο είναι παρόμοιο με το προηγούμενο. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα είναι ακόμη πιο σφιχτό λόγω των πολιτικών ευαισθησιών της ΑΦΕΤ αποφάσισε η ΑΦΕΤ ότι ήδη στις 16 Οκτωβρίου θα έχουμε το ψήφισμα για έγκριση. Θέλουν να το συζητήσουν τότε. Οπότε έχουμε μόνο μία δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε αν εργαστούμε ταχαίως και αν παρετηθούμε των μεταφράσεων σε όλες τις άλλες γλώσσες και δεχθούμε να συζητήσουμε με βάση το αγγλικό κείμενο. Αυτή θα ήταν η μόνη δυνατότητα χρονικά στις 6-7 Οκτωβρίου να το συζητήσουμε. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να δεχθείτε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον ε, εισηγητή μας τον κύριο Μόζαρ. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση που παρουσιάζω είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Για τη Γεωργία, την προηγούμενη. Και είναι και πολύ επίκαιρη στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης που κάναμε για την Ανατολική Γειτονία και την Ουκρανία και την κρίση στην Ουκρανία. Πολύ σύντομα να πω τα σημαντικότερα. Δεν θα αναφερθώ στις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν θα σας κουράσω, αλλά αν έχετε ερωτήσεις, επανέρχομαι. Η συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδαβία είναι πραγματική δυνατότητα σοβαρών αλλαγών για την Μολδαβία, όπως είπα και για τη Γεωργία. Δεν ε, σημαίνει δαπάνες για την Ένωση. Είναι μια βασική χειρονομία για μια ευρωπαϊκή χώρα που εύκολα μπορούμε να την κάνουμε. Στόχος συμφωνίας σύνδεσης είναι διτός η πολιτική σύνδεση και η οικονομική προσέγγιση των δύο πλευρών με βάση τις κοινέ μας αξίες και τους στενούς ιστορικούς δεσμούς. Πολλές φορές μιλάμε για κοινέ αξίες ε, και φαίνονται κενά λόγια, αλλά και για τη συζήτηση για την Ουκρανία που κάναμε τώρα, οι κοινέ λοιπόν αξίες αυτές που μοιράζομεθα, πρέπει να κατανοηθούν ως μεγάλη σημασίας. Ο κινητήρας της οικονομικής ε, προσέγγισης είναι αυτή η σε βάθος και σφαιρική Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου, DCFTA, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει προσέγγιση των προδιαγραφών σε μεγάλο βαθμό, θα εγκρίνουν λοιπόν και θα εφαρμόσουν τις ε, προδιαγραφές της Ένωσης σε πολλές από τις διαδικασίες παραγωγής τους και ο δεύτερος πυλώνας είναι η απελευθέρωση των αγορών. Η Μολδαβία είναι σε μεγάλο βαθμό γεωργική οικονομία, 36% του ΑΕΠ, τεράστιο, είναι γεωργικό, 27,5% της απασχόλησης στη γεωργία και 41% των εξαγωγών το 2011 που είναι τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία είναι γεωργικά προϊόντα. Οπότε κάνουμε φιλόδοξες παραχωρήσεις στο γεωργικό τομέα. Είναι βασικές για αυτή τη συμφωνία σύνδεσης και για τον DCFTA αυτό καθεαυτό. Οι παραχωρήσεις που κάνει η Ένωση είναι πολύ γενναιόδορες, πλήρη απελευθέρωση με την εξαίρεση έξι ευαισθητών προϊόντων, αν θέλετε λεπτομέρειε τι λέω. Ανάμεσα σε αυτά είναι το σκόρδο. Για τα φρούτα και λαχανικά, που είναι τμήμα τη συμφωνία. ad valorem και, συγκεκριμένα ε, είναι ε, χωρίς δασμούς οι εισαγωγές. για να αποφύγουμε ενδεχόμενο απατών από διάφορους εκεί στις ε, πρώην σοβιετικές περιοχές με κανόνες προέλευσης. Έχουμε ένα μηχανισμό για να αντιμετωπίζουμε τις προσπάθειες ε, παρεκκλήσεων ε, της διαδικασίας προέλευσης. Εάν φτάσουμε σε ένα κάποιο κατόφλι εισαγωγών, που να σημαίνουν ότι μάλλον οι εισαγωγές οι επιπλέον δεν είναι από τη Μολδαβία αλλά από άλλες χώρες, τότε υπάρχει ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης κόδων κινδύνου και μπορούμε να ζητήσουμε από τις μολδαβικές αρχές ότι αυτά τα προϊόντα όντως είναι μολδαβικά. Αλλά αυτά δεν είναι κρυφή φραγμή ή αν διαπιστώσουμε λοιπόν ότι αυξάνεται η παραγωγή της Μολδαβίας σε ένα προϊόν θα μπορούν να συνεχιστούν. Και η Μολδαβία έκαναν παραχωρήσει. Ουσιώδης βαθμός φιλευθεροποίησης εξαιρούνται λιγότερο από 100 γραμμές και για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα Υπάρχουν δυνατότητες ε, αντιμετώπισης. Μετά από τρία χρόνια θα γίνει μια κοινή προσπάθεια αναθεώρησης της συμφωνίας, ιδιαίτερα για τα TIQs. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν θα ξαναδούμε. Πρόσβαση στην αγορά, πλήρης απελευθέρωση και από τις δύο πλευρές, μόνο σταδιακό άνοιγμα των αγορών για μερικά ευαίσθητα προϊόντα, ευαίσθητα για την Μολδαβία. Ήδη ο βιομηχανικός τομέας ε, έχει μια ενδιαφέρουσα αντίδραση για την ε, εκ νέου βιομηχάνηση της ε, Μολδαβίας. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν εισαγωγικοί δασμοί για την εισαγωγή εξοπλισμού για τον τομέα των ανανεωσίμων και αυτό ήδη έχει οδηγήσει τους ε, βιομηχάνους εκεί να τονίζουν ότι θέλουν να αναπτύξουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Μολδαβία. Η πρόσβαση λοιπόν στην αγορά της Ένωσης για τη Μολδαβία βοηθάει την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης θα γίνει ευθυγράμμιση πολλών προδιαγραφών και κανόνων με τους δικούς μας. Η Μολδαβία θα ευθυγραμμίσει τους τεχνικούς της ε, κανόνες για τις υποδομές, για τα υγειονομικά και φυτο τα τελωνία από πλευράς πρακτικών και κανόνων και κανονισμών για να αποφύγουμε και τις απάτες και για τους λοιπόν ε, κανόνες προέλευσης η Μολδαβία θα ευθυγραμμίσει την νομοθεσία της για τα οικονομικά, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα ταχυδρομικές υπηρεσίες, τη χορήγηση αδειών, για να μην υπάρχουν ε, αυθαίρετες χορηγήσεις ε, αδειών σε διάφορους. Βέβαια κυρίως στη Μολδαβία είναι πρόβλημα αυτό. Δημόσιες προμήθειες, ε, πολύ θεαματικό, πλήρης αμοιβαία πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες προμήθεια, στη Μολδαβία θα ευθυγραμμιστούν με τους δικούς μας για να αποφύγουμε τη διαφθορά και την προσπάθεια ε, εισοδήματο που γίνεται στην ε, Μολδαβία. Όλα αυτά θα έχουν ε, επιπτώσει ε, στην οικονομική και πολιτική ελίτ όταν γίνονται όλα με βάση τους κανόνε και τη διαφάνεια οι πόροι δεν απομιζούνται, χρησιμοποιούνται σωστά. Είναι λοιπόν σημαντική η επίδραση στην ε, μεταλλαγή ολόκληρης της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Για την βιώσιμη ανάπτυξη συμφωνήσαμε σε πολύ γενναιόδορες ε, παραχωρήσεις. Οι κανόνες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασίας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας περιλαμβάνονται. Η Μολδαβία θα έχει μεγάλο κόστος οικονομικό να πληρώσει θα υπάρξει μεγάλη πίεση στην κοινωνία για να ευθυγραμμιστεί. Είναι όμως επένδυση στο μέλλον. Πρέπει όμως να γίνει και πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι δέχονται όλες αυτές τις δεσμεύσεις για να προσαρμοστούν και εμείς θα τους δώσουμε τις αναγκαίες οικονομικές και τεχνικές ε, προδιαγραφές, ε, ε, βοήθειες για να το κάνουν. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ θετικέ για την Μολδαβία. Μακροπρόθεσμα 5,4% αύξηση του ΑΕΠ προβλέπουμε λόγω αυτής της προσαρμογή, λόγω της συμφωνίας σύνδεση. Για τις επιχειρήσεις μα η αγορά θα είναι πιο σταθερή, προβλέψιμη και λίγα ακόμα για τις πολιτικές επιπτώσεις. δεν ε, στρέφεται κατά ή ουδήποτε. Είναι ελεύθερες επιλογές ελευθέρων συμβαλωμένων. Και όποιος ε, προσπαθεί να το δει διαφορετικά και θεωρεί ότι είναι συνωμοσία, δεν καταλαβαίνει τις αξίες μας. Επιμένω λοιπόν και σε αυτή την πλευρά. Γιατί ξεβλέπουμε ότι πολλοί ε, επιτίθενται κατά της ελευθερίας όπως στην Ουκρανία. Δεν θα κοστίσει λοιπόν πολλά, μόνο ωφέλει για την Ένωση. Έχει να κάνει βέβαια και με τις διαφορές ε, κλίμακας ε, μεταξύ Ένωσης και Μολδαβίας. Ε, είναι μικρή η Μολδαβία, μικρή επίπτωση λοιπόν στην Ένωση, αλλά θα είναι τεράστια επίπτωση στη μολδαβική οικονομία. Έχουμε λοιπόν μια δομή κινήτρων ούτως ώστε να υπάρξει μεταρρύθμιση του πολιτικού και θεσμικού πλαισίου σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε αυτή την συμφωνία και να δώσουμε την σύμφωνη γνώμη που θα προτείνει η ΑΦΕΤ στην Ολομέλεια για τη Συμφωνία Σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Λαντσμπέργης. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ ονόματος του κύριου Βίνκλερ. Η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μολδαβίας έχει στόχο να επιταγίνει την ευάθυνση και τη σύσφυξη των σχέσεών μας σε όλα τα επίπεδα ε, και σταδιακά θα ενταχθεί σε επιλεγμένους τομείς στην αγορά ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων στο DCFTA. Τους περασμένους μήνες ε, δεσμευτήκαμε και ε, για μια γρήγορη σύμφωνα με το Κοινοβουλίο και καλέσαμε τα κράτη-μέλη αμελητή να κυρώσουν τη συμφωνία. Δεδομένων των παρουσών πολιτικών συνδικών είναι ακόμα πιο επίγουσα η κατάσταση. Στην ΑΦΕΤ θυμίζω ότι αποφασίστηκε ε, χωρίς καμία αντίρρηση να επιταχυνθεί η διαδικασία έτσι ώστε να έρθει στην Ολομέλεια στις 12 και 13 Νοεμβρίου λίγες μέρες πριν τις γενικές εκλογές του τέλους Νοεμβρίου στη Μολδαβία. Ζητούμε λοιπόν ε, μία σύντομη και ταχεία έγκριση της ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ, ο Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς και καταρχήν πιστεύω ότι έχουμε ε, το ίδιο πλαίσιο με την Ουκρανία. Είναι μια χώρα σε μετάβαση που έχει να αντιμετωπίσει την εξή κατάσταση. Τώρα ξεχρονίζω την οικονομία μου, με ποιον εταίρο θα το κάνω. Ε, και αυτό ισχύει και για τη δημοκρατία της Μολδαβίας και ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση της γνωμοδότησης και της εξηγήσει που μας έδωσε. Τονίζει λοιπόν, ετώνησε δύο-τρεις φορές αν δεν απατώμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρωτώ ποιος ωφελείται από αυτή τη συμφωνία. Γνωρίζοντας ότι 90% της μολδαβικής οικονομίας προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τους ρωτήσατε γιατί αντίκτυπο θα έχουν αυτές οι συμφωνίες και εφαρμογή τους στη δική τους οικονομική κατάσταση και της χώρας. Όπως είπατε είναι μια περίπλοκη διαδικασία μετάβασης αυτή που διέρχεται η χώρα. 90 ή 80% δεν έχει σημασία. Ε, εστιάζεται κυρίως στη γεωργική παραγωγή. Και τίθεται ήδη σε ισχύ και εν αυτών η Ρωσική ε, Ομοσπονδία έχει αυξήσει τους δασμούς. Δηλαδή, και πάλι μπαίνουμε σε αυτό το θέμα. Ποια θα είναι η μελλοντική σχέση σε αυτό το τρίγωνο ε, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση Μολδαβία ε, και ε, Ρωσική Ομοσπονδία στη ροή των αγαθών. Και είναι σημαντικό αυτό για τη Γεωργία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμη να δώσει στη Μολδαβία πρόσβαση στις αγορές της τώρα αμέσως ε, μετά την 1η Σεπτεμβρίου σε αυτό το διάστημα που διανύουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα που συνδέεται με την ίδια τη σταθερότητα της χώρας. Ξέρουμε ότι έχει βουλευτικές εκλογές, γι' αυτό εμείς είμαστε κατά της επιτάχυνσης της διαδικασίας. Και με φαίνει αυτό στο εξή ερώτημα. Πιστεύουμε εμείς ότι στέλνουμε το σωστό μήνυμα στην κοινωνία της Μολδαβίας. Βοηθούμε και τη συζήτηση και την κοινωνία την ίδια να επιλέξει μια προοπτική για το μέλλον της και να επιλέξει, μάλλον να, να αποδεχτεί ότι είναι δύσκολη αυτή η μεταβατική περίοδος ή μήπως κινδυνεύουμε να οδηγήσουμε σε διχασμό ε, την κοινωνία. Ξέρετε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι κατά αυτής της διαδικασίας ενώ το Κομμουνιστικό είναι υπέρ. Δηλαδή είναι μεγάλη η σύγκρουση εκεί. Και γίνεται μια ολόκληρη κοινωνική συζήτηση Και λάβουμε δε υπόψη ότι ε, το μηνιαίο εισόδημα ενός μισθωτού, ενός εργαζομένου στη Μολδαβία είναι 100 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό. Αν έχουν εύκολη πρόσβαση οι ευρωπαϊκές εταιρείες και πιέζουν στον ανταγωνισμό με τις μολδαδικές. θα υπάρχει δυνατότητα για τις μορταβικές εταιρείε να είναι σε γνήσιο πραγματικό ανταγωνισμό με τις ε, επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια τελευταία ερώτηση, αναφερθήκατε στις δημόσιες προμήθειες κτλ. Αυτό τι θα σημάνει. Θα ε, κλείσουν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, κοινοφελίες ή θα παραμείνουν ως το παρόν καθεστώς. Δηλαδή μπορεί να χαθούν θέσεις εργασίες και όλη αυτή είναι μια συζήτηση προς τα που θα στραφεί η χώρα τελικά, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ευχαριστώ, Ιγνάσιο. Uh, yes, thank you very much, Ευχαριστώ. Ευχαρίστως να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Σόλτς. Να πω όμως ότι ε, η Κομισιόν καλωσορίζει ε, και επιθυμεί την γρήγορη επικύρωση αυτής της συμφωνίας ε, γιατί είναι ένας σημαντικός εταίρος και έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά την ταχεία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ε, για την περίπτωση της Μολδαβίας ε, στην ε, διάμεση εφαρμογή, την προσωρινή εφαρμογή είχαμε ήδη το ποσοστό του 45% όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και βεβαίως έχουμε, έχουμε θέσει λειτουργία το μηχανισμό αυτόν ο οποίος αποτρέπει την παράκαμψη των διαδικασιών. Πέρα από αυτό υπάρχει πλήρης πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ε, για τις εξαγωγές μολδαβικών προϊόντων. Επίσης ε, πρέπει να σας πω ότι από πλευρά της Κομισιόν έχουν ληφθεί και γίνει σεβαστή υπόψη όλοι, όλες οι ιδιαιτερότητες ε, και όλες οι ευαισθησίες της Μολδαβίας και όσον αφορά την ευθυγράμμιση πρέπει να πω ότι επίσης ε, έχουμε συμφωνήσει με τις προτεραιότητες τις οποίες η ίδια η Μολδαβία έχει καθορίσει έτσι ώστε να υπάρξει βαθμιαία προσέγγιση και ευθυγράμμιση μάλλον με το ε, κοινοτικό ε, κεκτημένο. Όσον αφορά τώρα τις δημόσιες προμήθειες, ε, οι δεσμεύσεις ε, που έχουν αναλυφθεί είναι, οδηγούν προς την ευθυγράμμιση ε, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα και δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα, άρα δεν υπάρχει λόγος προβληματισμού επ' αυτού. Είναι γεγονός ότι η ε, ε, Μολδαβία έχει υποστεί σημαντική πίεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία η οποία αποφάσισε να μην ε, συνεχίσει την εφαρμογή των προτιμησιακών καθεστώτων για την Μολδαβία έστω και αν είναι μικρό το ποσοστό της ε, Μολδοβίας, ε, παρόλα αυτά αποφάσισαν να μην ε, συνεχίσουν το προτιμησιακό καθεστώ και επίσης για υποτιθέμενους λόγους έχουν προχωρήσει και σε κάποιες ακυρώσεις όσον αφορά την Μολδαβία. Γι' αυτό λοιπόν αυτό αποτελεί ένα λόγο παραπάνω έτσι το Κοινοβούλιο γρήγορα να κυρώσει την συμφωνία. και αργότερα θα συζητήσουμε και άλλα θέματα όταν προκύψουν αυτά σχετικά με επιπλέον ανοίγματα προς τη Μολδαβία. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής για μία ακόμη φορά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Πολύ καλές ερωτήσεις σας. Μερικές είναι και φιλοσοφικού χαρακτήρα θέλει. Για τις ε, δημόσιες κοινοφελείς υπηρεσίες νομίζω απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο πολύ ξεκάθαρο. Τώρα, αν θα υπάρξουν δυνατότητες για γνήσιο ανταγωνισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Μολδαβίας. Μα μπορεί να σας φανεί αυτό στερεότυπο, αλλά έχοντας πρόσβαση στην υπαριθμό ένα αγορά του κόσμου, με χαμηλούς μισθούς, στην αρχή της ανάπτυξης ενός οικονομικού κύκλου είναι ευκαιρία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εάν νομικά στην αρχή υιοθετήσει ε, τα πρότυπα, ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά δημιουργούνται και διανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες για τους επενδυτές. Ε, μπορεί να ασκήσει κάποια πίεση αυτό στους μισθούς, οι νέες τεχνολογίες που έρχονται στη χώρα. Ένας ολόκληρος κόσμος όμως ευκαιριών διανοίγεται για καινοτομία και πρόοδο ενδεχομένω. είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης στραμμένο προς εξαγωγές, εξωστρεφές και στις ελεύθερες συναλλαγές. Και... Μακροπρόθεσμα θα είναι αυτό πιο ευνοϊκό για ε, τις ευρωπαϊκές ή για τις μολδαβικές επιχειρήσεις. Ε, νομίζω ότι και οι ε, μολαβικές επιχειρήσεις το επιθυμούν. Κοιτάξτε, η Ρωσία δεν είναι ανταγωνιστική. Ε, βασίζεται πάρα πολύ στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για την ανάπτυξή της. Ενώ η πραγματική κοινωνική ανταγωνιστικότητα με οικονομικούς όρους είναι ασθενής. Δηλαδή, εάν η Μολδαβία προσδεθεί προς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι καταδικασμένη σε μια επανάπτυξη διαρκείας. Εάν προσδεθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρξει στην αρχή ένα, σοκ στην αρχή για την προσαρμογή της, αλλά θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στη συνέχεια. Πέρα από τα στερεότυπα. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ευθυγραμμιστεί νομοθετικά και κανονιστικά προς αυτή την αγορά. Ε, είναι υπέρ της, είναι του... <laughs> Δεν ξέρω, είναι μια ε, ίσως απλή απάντηση για τη μακροπρόθεσμη προοπτική που διανοίγεται. Αυτά. Ευχαριστώ Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω καμιά αντίρρηση με το πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα και τι τροπολογίε στα αγγλικά. 29 λοιπόν του μηνό 6 το απόγευμα, λήξη προθεσμίας, αν συμφωνείτε. Και εφόσον συμφωνείτε, είπαμε οι τροπολογίε ε, θα είναι είτε για έγκριση είτε για απόρριψη. Ναι ή όχι, αλλά υπάρχει και το συνοδευτικό ψήφισμα βεβαίω. Ε, και οι ε, τροπολογίε θα συζητηθούν εδώ στι 6 Οκτωβρίου, ενώ στι 7 του μηνό Οκτωβρίου θα ψηφιστούν. Ε, όποιος ε, θέλει να συνεχίσει να ακούει τον Ιγνάσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθεί ακρόαση για τι κυρώσει από τη Ρωσία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι ένα από του ομιλητέ. Η συνάδελφο Σαράντσοβα ε, το έχει διοργανώσει. Ε, αν θέλετε κατά τη διάρκεια του διαλύματο, αν δεν τον ακούσετε αρκετά στην Επιτροπή μα να πάτε να τον ακούσετε και εκεί. Ευχαριστώ. Λήξη τη συνεδρίαση και σε λίγο θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ. Ευχαριστώ πολύ.